λόγια, ακριβώς επειδή έχουμε καθυστερήσει πολύ, να σας ενημερώσω για το πώς ε, θα διεξαχθεί αυτή η ώρα των ερωτήσεων. Και σας θέρμα παρακαλώ να δώσετε λίγη προσοχή και οι επίτροποι που θα κληθούν να απαντήσουν. Ως συμπληρωματικές ερωτήσεις θα ακούμε μόνο τις ερωτήσεις των συντακτών των ερωτήσεων, δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε και άλλες συμπληρωματικές ερωτήσεις και θέλω να διεκπαιρεώσουμε όσο δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις γίνεται και θα ήθελα να θερμοπαρακαλέσω και τους επιτρόπους που απαντούν να μην διαβάζουν μακρινάρια. Μας ενδιαφέρουν συνοπτικές και περιστατωμένες απαντήσεις ώστε να δημιουργείται ένας γνήσιος διάλογος και με τον συντάκτη της ερώτησης. Ο κύριος Λάιτφριντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να ομολογήσω ότι όσον αφορά αυτά που είπατε σχετικά ε, με την καθυστέρηση, ε, τα κατανοώ, αλλά θα ήθελα να λάβετε υπόψη και το εξή. Αυτοί που θέλουν να κάνουν τις ερωτήσεις τους, ε, αυτοί δεν φταίνε που καθυστερήσατε τόσο πολύ και εγώ έχω ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Δηλαδή, στο σημείο υπαριθμών 2, εγώ υποβάλλω μια ερώτηση προς το Συμβούλιο και ε, την είχα υποβάλει στην ώρα του Συμβουλίου και δεν μπόρεσα να την κάνω. Αυτό πολύ, με δυσαρέστησε, πολύ με δυσαρέστησε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω ε, ίσως ε, γι' αυτό το ένα και μοναδικό σημείο να αναθεωρήσετε λιγάκι αυτά που είπατε, να κάνετε μια εξαίρεση. Δυστυχώς ε, οι συνθήκες με υποχρεώνουν να είμαι τόσο αυστηρή και Λοιπόν, λυπούμε ειλικρινά για τους συντάκτε των ερωτήσεων, αλλά το, αυτό που ενδιαφέρει είναι να απαντήσουμε όσο, το δυνατόν περισσότερες ερωτήσει γίνεται, δίνοντας δικαίωμα στην πληρωματική ερώτηση μόνο στο συντάκτη της ερώτησης. Ξέρετε ότι δεν μου αρέσει και πολύ αυτή η κατάσταση, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να εξυγχρονίσουμε την ώρα των ερωτήσεων και να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αλλά ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Μακάρι να έρθει το συντομότερο δυνατόν. Η πρώτη ερώτηση είναι η ερώτηση Μπλίνκεβιτσούτε, αφορά την οδηγία πλαίσιο σχετικά με το ελάχιστο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απευθύνεται προς τον Επίτροπο Άντορ. Ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη και ευρωβουλευτές. Πολλές φορές λέμε ότι η κοινωνίε κρίνονται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα ασθενέστερα μέλη του. Γιατί αν δεν ε, βοηθήσουμε του αναξιοποιηθεί και αυτού ε, που έχουν περισσότερη ανάγκη, θα του περιθωριοποιήσουμε ακόμη περισσότερο αντί να προσπαθήσουμε να του εντάξουμε στην κοινωνία και να του φέρουμε στην αγορά εργασία. Πιστεύουμε ότι εκτό ότι ε, είναι σταθεροποιητέ, τα συστήματα ελάχιστων εισοδημάτων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο γιατί προστατεύουν του πλέον ευάλωτου από πιο ελεύθερη αποτελέσματα τη κρίση χορηγώντας κάποιε ασφαλιστικές ε, δικλείδε και δίκτυα ασφαλεία. Και μάλιστα τα αποτελέσματα του Συμβουλίου της 17 η Σεπτεμβρίου του 2008 για τις αρχές αποτελεσματικής καταπολέμησης της φτώχεια, δείχνουν τη σημασία που έχει πρόσβαση σε κατάλληλου πόρους αλλά και σε ποιοτικέ υπηρεσίες και αγορέ εργασιών που θα ε, συμπεριλαμβάνουν και δεν θα αποκλείουν. Καλούμε τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των, ιδιωτών, των πολιτών σε πόρους και κοινωνική παροχή, προκειμένου να ε, μπορέσουν να ζούμε αξιοπρέπεια. Και αυτό είναι τμήμα της ε, προσπάθειας καταπολέμησης τη κοινωνική περιθωριοποίησης. Ε, οι προτάσει μας ε, είναι ένα βήμα προ σωστή κατεύθυνση, ιδιαίτερα στα πλαίσια της κρίσης. Αλλά φυσικά χρειάζομαστε και νέα μέτρα για να εφαρμόσουμε πλήρως και αποτελεσματικά την μεταρρύθμιση υπέρ της κοινωνικής ένταξης. Είναι πολύ σημαντικό και το 2012 σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της κοινή αρχής για την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία που στηρίζονται και στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελάχιστου εισοδήματο. Προτείνουμε δράσεις που ανάλογα με την αξιολόγηση και τα αποτελέσματά της θα περιλάβουν και χρηματοοικονομικά μέσα για την ενεργό πραγματικά συμμετοχή στην κοινωνία. Κύριε Βλυνκεβιτσούτε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο για την απάντηση. Βέβαια, δεν νομίζω ότι απαντήσατε ακριβώς την ερώτηση, κύριε Επίτροπε, γιατί η ερώτησή μου είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει μια οδηγία για την εξασφάλιση του ελάχιστου εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Πέρυσι, που ήταν το έτος της καταπολέμησης της φτώχειας, διαπιστώσαμε ότι η φτώχεια αντί να μειωθεί, αυξήθηκε. Και η δεύτερη μου ερώτηση είναι τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ηλικιωμένου. Γιατί και οι ηλικιωμένοι πλήττονται ιδιαίτερως από την ε, φτώχεια. Πρόκειται να προτείνετε κάποια ομοιόμορφα κριτήρια για τις συντάξεις. Είπαμε για το ελάχιστο εισόδημα και τους ελάχιστους μισθούς, αλλά αυτά είναι εθνικές αρμοδιότητες. Εδώ ισχύει η αρχή της επικουρικότητας. Συγγνώμη κύριε Επίτροπε. Υπάρχει ένα πρόβλημα διερμηνίας, λέει η Πρόεδρος. Από τα αγγλικά ακούγεται άλλη γλώσσα. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Μπορείτε να ξαναρχίσετε κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρα ε, του ελάχιστου εισοδήματο και του ελάχιστου μισθού, αλλά αυτό αποτελεί εθνική αρμοδιότητα και εθνική ευθύνη. Γιατί εδώ ισχύει η αρχή της επικουρικότητας που υπερισχύει. Βέβαια, σε περίοδο κρίσης θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στους πιο ευάλωτους πολίτες της κοινωνίας και στις πιο ευάλωτες ομάδες και ιδιαίτερα αυτούς που δεν έχουν εισόδημα, τους απόρους ή τους άνεργους. Επίσης θα πρέπει να θαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν κάθε δυνατό μέσο για να αποτρέψουν την διολίσθηση των πολιτών στη φτώχεια. Αλλά το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτό είναι πολύ περιορισμένο, παρόλο που και η πολιτική έκκληση έχει τη σημασία της. Σε ό,τι αφορά τη φτώχεια για τους ηλικιωμένους, το θέμα αυτό είναι πολύ περίπλοκο και έχει σχέση με την απασχόληση, με τις κοινωνικές υπηρεσίες, με την κοινωνική πρόνοια και προστασία και σχετίζεται και με την εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, ενεργό και δραστήρια γύρανση και αφορά και την προστασία της υγείας, ε, τη διαβιοκατάρτιση, κατάρτιση, γιατί πιστεύουμε ότι η μεγαλύτερη πρόοδος που μπορούμε να, να επιτελέσουμε για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων είναι ε, ενισχύοντας τη συνεργασία τους στην αγορά εργασίας και με κάποιες συμπληρωματικές πολιτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Περνάμε στη δεύτερη τώρα ερώτηση που είναι ερώτηση της κυρίας Σιλβάνα Κοχμερίν για τις λεπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Η ερώτηση αυτή απευθύνεται στον Επίτροπο Έτιγκερ. präsidentin frau abgeordnete koch marin meine damen und herren abgeordnete! κυρία ε, βουλευτά είναι γνωστή αυτή η έκθεση ε, της αρμόδιας υπηρεσίας και επίσης ε, εξετάστηκε το θέμα σε βάθος. Η άποψη, η απόφαση που λήφθη είναι εξής. Λόγω της απόφασης του Συμβουλίου και κατόπιν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και του Συμβουλίου Ενέργειας, δηλαδή στο Κοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη έγιναν διαβουλεύσεις και η Κομισιόν το 2009 στη δική της ε, την πρόταση ε, έκανε τη δική συμπρόταση σε έναν κανονισμό eco-design όπου αναφέρεται η σταδιακή μετάβαση από τους ε, συμβατικούς λαμπτήρες σε ε, λαμπτήρες που χρησιμοποιούν οικονομικά την ενέργεια. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι στην ευρωπαϊκή αγορά για λαμπτήρες μπορεί να υπάρξει και υπήρξε εξοικονόμηση μέχρι 20 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες. Αυτό σημαίνει 5 μέχρι 10 δισεκατομμύρια ευρώ εξοικονόμηση κόστους ενέργειας. Ε, με την οδηγία αυτή λάβαμε διάφορα μέτρα και το Σεπτέμβρη του περασμένου έτους ε, προβήκαμε σε περαιτέρω μείωση για να αντιμετωπίσουμε δυνάμει κινδύνους και να τους ελαχιστοποιήσουμε περαιτέρω έκθεση λοιπόν του, ε, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος μας οδήγησε να παρακαλέσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες να τοποθετηθούν και μετά από τον έλεγχο της επιστημονικής βιβλιογραφίας η αρμόδια αυτή επιστημονική επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ε, ο κίνδυνος για την υγεία ε, στην περίπτωση που σπάσουν αυτοί οι λαμπτήρες ε, δεν υπάρχει κίνδυνο για την υγεία, είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Οι μελέτες αυτές βασίζονται ε, σε έρευνες που έγιναν με ενήλικες. Βεβαίως τα παιδιά πρέπει να εξεταστούν ως ειδική περίπτωση και γι' αυτό λοιπόν ήρθαμε πάλι σε επαφή με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος ζητώντας το συντομότερο δυνατόν να μας παρουσιάσουν τα αποτελέσματα και για τα παιδιά Παρακολουθούμε την ε, κατάσταση εκ του ε, Έχουμε απευθυνθεί, όπως σας είπα, στο ομοσπονδιακό, στην Ομοσπονδιακή Υφτή Υπηρεσία, έτσι ώστε τα στοιχεία να μας κατατεθούν και να αξιολογηθούν το συντομότερο δυνατόν. Βεβαίως, ε, επειδή πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, εμείς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο κανονισμός αυτός ε, θα συνεχίσει να ισχύει και αν όμως εντωμεταξύ αποκτήσουμε διαφορετικά συμπεράσματα που οδηγούν σε διαφορετικά ε, μέτρα, θα ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο. Η κυρία Κοχμερίν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ κύριε Οτιγκέρ, κύριε Επίτροπε, πολύ καλά όλα αυτά που μας είπατε, που αναθέσατε εκ νέου το θέμα στην Επιστημονική Επιτροπή. Πάντως το θέμα παραμένει. Πώς είναι δυνατόν να εξηγήσει κανείς τους πολίτες της Ευρώπης ότι ε, τελικά στα παιδιά τους υπάρχει κάτι το οποίο προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι επικίνδυνο για τα ίδια τους τα παιδιά. Ε, το πρόβλημα υπάρχει και στην Αυστρία. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι ότι υπάρχει κάτι το επικίνδυνο. Ε, εσείς ε, βέβαια δεν το υπερασπιστήκατε και γι' αυτό δεν χρειάζεται να φοβάστε ότι ενδεχομένως θα εκτεθείτε. Αλλά θα ήθελα πραγματικά να λάβετε για άλλη μια φορά υπόψη σας όλα αυτά που αναφέρθηκαν σχετικά με τους κινδύνους που να υπάρχουν στα νοικοκυριά ο Επίτροπος. Ε, θα ήθελα να σας ε, επισημάνω το εξής. Στην αγορά και μετά την αλλαγή με τους λαμπτήρες ακόμα και αν πράξουν και περαιτέρω αλλαγέ, θα εξακολουθούν να υπάρχουν λαμπτήρες που δεν θα είναι επικίνδυνοι. Εσείς ε, αναφέρεστε στις CFL, στους CFL λαμπτήρες Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα ήθελα να σας ε, ενημερώσω για τη δική μας ε, τη δουλειά, τη δουλειά που κάναμε σχετικά με την οδηγία designer. Ε, Θελήσαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες για τους προβολείς LED και για τους προβολείς με αλογόνο. Όλα αυτά βέβαια έγιναν στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας. Ε, θελήσαμε να αποκλείσουμε οποιαδήποτε μορφή κινδύνου. Ε, και αν θέλετε πολύ ευχαρίστω να επανεξετάσουμε το θέμα σε βάθος. Ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια ε, του, των ερωτήσεων δεν δεχόμεθα μπλε κάρτες. Καλό ήταν αυτό που δοκιμάσατε, αλλά δεν έπιασε. Επόμενη ερώτηση λοιπόν αφορά ε, τα ε, θύματα, δέσμη μέτρων για τα δικαιώματα των θυμάτων. Ε, η κυρία Ρέντιν θα απαντήσει. Do I have the floor? Πρόεδρε, μου δίνετε το λόγο, λέει η κυρία Ρέντινγκ. Μάλιστα. Γνωρίζετε ότι πάνω από 30 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δηλώνουν ε, κάθε χρόνο ότι είναι θύματα εγκληματικών ενεργειών. Και βεβαίως θα πρέπει να βεβαιώσουμε ε, τη δυνατότητα των θυμάτων να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματά τους και να ε, απολαμβάνουν τις προστασίες που χρειάζεται. Είναι προτεραιότητα αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα επευκαιρία να ξάρω το θάρρος της κυρίας Χιούτς που αγωνίζεται ε, για ε, τη μεγαλύτερη υποστήριξη των θυμάτων σε όλη την Ευρώπη και το σένος της και η αποφασιστικότητά της θα πρέπει να είναι για μας όλους παράδειγμα για να ενισχύουμε τα δικαιώματα των πολιτών και των θυμάτων για να έχουν και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ένωμη τάξη μας οι πολίτες. Χρειαζόμαστε αμοιβαία εμπιστοσύνη για να ε, ξέρουν οι πολίτες ότι προστατεύονται και αναγνωρίζονται τα δικαιώματά τους όχι μόνο στην επικράτεια της χώρας τους αλλά και ε, διασυνοριακά. Επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε να μην λησμονούνται τα θύματα από το δικαστικό σύστημά μας και το νομοθετικό. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει ένα συνολικό πακέτο για τα θύματα για να αντιμετωπίσει την ποιότητα της υποστήριξης που ε, δέχονται τα ε, θύματα ε, μετά την εγκληματική ενέργεια και κατά τη διάρκεια της δίωξης και της όλης δικαστικής διαδικασίας ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης ή την εθνικότητά τους. Οι προτάσεις μας θα συμπεριλαμβάνουν την αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς προς τα θύματα για να μην υφίστανται και περαιτέρω ζημία και βλάβη κατά τη διάρκεια των ε, δικαστικών διαδικαστικών ε, για να μην είναι διπλή η θυματοποίησή τους. Τι θα είναι αυτά τα μέτρα. Οριζόντια οδηγία ε, για τη θέση των θυμάτων σε ποινικέ δίκες ε, με δικαιώματα που να ε, μπορούν να διεκδικηθούν και να επιβληθούν εύκολες ε, υπηρεσίες υποστήριξη θυμάτων, το δικαίωμα της διερμηνίας κατά τη διάρκεια των καταθέσεων και δυνατότητα χωριστών θουσών αναμονής για τα θύματα στα νέα κτίρια που χτίζονται των δικαστηρίων ε, και ε, τα λοιπά. Στη συνέχεια θα προτείνω ένα κανονισμό για ε, μέτρα προστασίας στο αστικό δίκαιο. Δηλαδή οποιοδήποτε θύμα κινδυνεύει και χρειάζεται να μπει ένα σύστημα προστασίας σε ένα κράτος μέλος να μπορεί να απολαμβάνει αυτής της προστασίας όταν ταξιδεύει σε άλλο κρατός μέλος. Το μέσο αυτό θα συμπληρωθεί από ένα άλλο μέτρο για αμοιβαία αναγνώριση μέτρων ε, ε, στο ποινικό δίκαιο. Επίσης θα λάβουμε και μέτρα και πολλά μη νομοθετικού χαρακτήρα για να βεβαιωθούμε ότι θα ε, εκτελούνται σωστά η νομοθεσία και θα προτείνουμε και μέτρα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων για να είναι προτεραιότητα παντού και να παραμείνει και τα επόμενα έτη αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μωράες. Κύριε Επίτροπε, όπως γνωρίζετε, ήρθαμε στο γραφείο σας την περασμένη εβδομάδα με τη Μάγκη Χιούς, ε, που είναι μία από τους πολλούς χιλιάδες ε, που έπεσαν θύματα εγκληματικών ενεργειών. Και πρέπει να σας πω ότι μετά τις επαφές που είχαμε στο γραφείο σας χαρήκαμε πάρα πολύ για τα μέτρα αυτά που θα προσφέρουν εμπιστοσύνη και προστιθέμενη αξία στα θύματα που χρειάζονται υποστήριξη. Ε, η Μάγκη Χιούς και πολλά άλλα θύματα εγκληματικών ενεργειών μας είπαν ότι τα μέτρα που προτείνεται είναι ωραία και καλά, αλλά αυτό που θέλουν να δουν εκείνοι είναι μια συγκέντρωση στην παροχή βοήθειας. Ε, ας πούμε να υπάρχει ένα γραφείο, μια υπηρεσία στην οποία να αποτείνονται ε, με ευκολία ε, να υπάρχουν πρόσωπα που να τους βοηθούν στα νοσοκομεία, στα αστυνομικά τμήματα, στα δικαστήρια. Αυτό ζητούν και μέχρι τώρα αυτό δεν τους παρέχεται είναι πραγματικά μια έκκληση που απευθύνουν σε εσά για να αυξηθεί η πρόταση και η προστασία τους όσο γίνεται περισσότερο. Η Επίτροπος. Συμφωνώ πολύ με τον κύριο Βουλευτή. Τα θύματα ε, έχω την αίσθηση είναι λίγο απόντα μέχρι τώρα. Ε, διαβάζοντας ε, τη δικονομία ε, Βλέπω ότι δίνουμε μεγάλη προσοχή στο φερόμενο ως δράστη ε, ε, μιας αξιόπινης πράξης και ασχολούμαστε πολύ με την υπεράσπιση του κατηγορουμένου. Αυτό είναι κάτι που βεβαίως θα πρέπει να κάνουμε και καλά κάνουμε και το πράττουμε σε μια κοινωνία σαν τη δική μας που βασίζεται σε δικαιώματα. Αλλά πολλές φορές τα θύματα πέφτουν ε, για δεύτερη φορά σε αυτή την κατάσταση, οι θύματα, ε, όταν φτάνει η υπόθεση στην ακροματική διαδικασία στο δικαστήριο. Ε, γι' αυτό ε, το πακέτο αυτό για την προστασία των θυμάτων και τα δικαιώματά τους ελπίζω να αλλάξει όχι μόνο τους νόμους αλλά και τις νοοτροπίες. Παντού, δηλαδή, στα δικαστήρια μας, στα αστυνομικά μας τμήματα, στα νοσοκομεία, όπως είπε πολύ σωστά ο αξιότιμος βουλευτής, να έχουν ειδική φροντίδα τα θύματα. Και ξέρουμε ότι δεν ε, είναι η ίδια μεταχείριση που θα πρέπει να ε, τους επιφυλάσσουμε όπως με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Και αυτό να μην ισχύει μόνο στη δική τους χώρα αλλά και στις υπόλοιπες υπολογίζω στο Κοινοβούλιο να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει όσο γίνεται καλύτερη νομοθεσία σε αυτό το τομέα και στα στοιχεία της συναπόφασης ε, του πακέτου να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία στο Κοινοβούλιο έτσι ώστε να επιτευχθεί τελικά συμφωνία στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Περνάμε στην επόμενη ερώτηση της κυρίας Χάρκιν προς τον Επίτροπο Σεμέτα αφορά τις προτάσεις Επιτροπής σχετικά με μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των επιχειρήσεων. Ο Επιτροπός Σεμέτα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των επιχειρήσεων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έρει τους φραγμούς της ευρωπαϊκής αγοράς όπως φάνηκε από την ε, ε, μελέτη που πραγματοποιήθηκε. Επίσης, ε, ε, δημιουργεί η έλλειψή της ε, φραγμού στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η, η αποκλήση μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων πολλέ φορέ οδηγεί σε διπλή φορολόγηση, υπερβολική φορολόγηση των επιχειρήσεων. Όλο και περισσότερο οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει αντιμετωπίζουν τεράστιο γραφειοκρατικό άχθο και έχουν τεράστιο κόστο ε, με τη συμμόρφωση με τους κανόνες. Αυτό δημιουργεί αντικίνητρα σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητά τους και απάδει με την, με την πρόταση για το 2020. Θα πρέπει να προσφέρουμε ενιαίο πακέτο μέτρων για τις ε, επιχειρήσεις που θα διευκολύνουν τις ε, δραστηριότητές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοινή ενωπημένη βάση φορολογία των επιχειρήσεων θα εξεταστεί στις 16 Μαρτίου από, το, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύω ότι θα συμβάλλει στη βελτίωση του, επιπέ, του περιβάλλοντος και του κλίματος και για τις επιχειρήσεις και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Χάρκιν, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Έχω τρεις σύντομε ερωτήσεις συμπληρωματικά και ελπίζω να μπορέσετε να τι απαντήσετε η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των επιχειρήσεων θα είναι προαιρετική με βάση την πρότασή σας και υπό ποιες συνθήκες ε, τα τοπικά δικαστήρια μπορούν να χάσουν την ε, δικαιοδοσία τους για φορολογικά θέματα και ποιες θα είναι, αυτές οι... και ποιες είναι οι επιπτώσεις σε άλλα κράτη-μέλη. Φαντάζομαι υπάρχει και μία ανάλυση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ποιοι είναι κερδισμένοι και ποιοι χαμένοι από οικονομική άποψη ε, ανάλογα με την πρόταση που θα υιοθετήσει τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την ίσπραξη φόρου σε άλλο κράτος μέλος. Ο Επιτροπές θα είμαι και εδώ πολύ σύντομο σε ό,τι αφορά το κατά πόσο θα είναι προαιρετική ή υποχρεωτική η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογία των επιχειρήσεων. Θα είναι προαιρετική η βαση φορολογιας των επιχειρησεων θα είναι και θελής η βαση θα ειναι και η εφαρμογη της. Η πρότασή μας είναι για μια ε, εθελοντική τέτοια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των επιχειρήσεων και δυνατότητα των επιχειρήσεων να την εφαρμόσουν ή όχι. Σε ό,τι αφορά το ρόλο των ε, τοπικών δικαστηρίων και της δικαιοδοσίας τους και τι γίνεται με τον διακανονισμό των διαφορών, ποιος είναι ο ρόλος των τοπικών δικαστηρίων, η πρόταση για την κοινωνιοποιημένη βάση φορολογία των επιχειρήσεων δεν πρόκειται να επηρεάσει τους κανόνες δικαιοδοσίας και δοσηδικία των δικαστηρίων. Η κοινωνιοποιημένη βάση φορολογία των επιχειρήσεων είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούμε που και που θα μοιράζεται μεταξύ των των πωλήσεων, του εργατικού δυναμικού και των ε, περιουσιακών στοιχείων, των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης. Και θα λαμβάνει υπόψη το τζίρο και τον αριθμό των ε, εργαζομένων. Έγινε και μελέτη επιπτώσεων που θα δημοσιευθεί από κοινού με την πρότασή μας. Είμαι πεπισμένος πάντως ότι η πρόταση αυτή θα βοηθήσει και θα είναι επωφελής και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις γενικά και για τις ελλαδικές επιχειρήσεις ειδικά. Βλέπω λοιπόν ότι έρχονται κάποιοι στην αίθουσα αυτή ακριβώς επειδή έχουμε την ώρα των ερωτήσεων. Ε, τελικά δεν θα έχουμε και τόσο μεγάλη πίεση. Βέβαια, στόχος μας είναι να απαντήσουμε όσο το δυνατόν ε, περισσότερες ερωτήσεις. Είπα όμως στην αρχή ότι δεν θα δεχτούμε συμπληρωματικές ερωτήσεις, εκτός από εκείνους που έχουν υποβάλει ερωτήσεις. Τώρα, λοιπόν, να σας πω, ο στόχος μου είναι και εξαρτάται βέβαια σε κάποιο βαθμό από ε, το πόσο θα μιλήσουν οι Επιτροποί. Πριν από τις 9 παρατέταρτο, μέχρι τις 9 παρατέταρτο να εξετάσουμε τις ερωτήσεις Γένσεν Παπα-Νικολάου, Πόσελτ, Κικάου. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Η ερώτηση της κυρίας Γένσεν ε, προς ε, τον Επίτροπο Σεμέτα που αφορά την απαλλαγή από το ΦΠΑ για γεωργικά προϊόντα στη Ρουμανία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λόγω του ότι υπάρχουν απάτες με το ΦΠΑ ε, σε κάποιες περιπτώσεις γενικών προϊόντων, η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Μία λοιπόν από τις λύσεις που μπορούν να προκύψουν με αυτές τις ε, απάτες ε, καρουσέλ Έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα ε, που αφορά την εξαίρεση του ΦΠΑ ε, και το πρόγραμμα αυτό προβλέπει ότι ε, το ΦΠΑ δεν τον καταβάλει πλέον ο προμηθευτής αλλά ο αποδέκτης. Αυτή είναι η μόνη τροποποίηση στο καθεστώς που ισχύει όπου Κανονικά ο προμηθευτής καταβάλει ε, τον φόρο, ο αποδέκτης ε, τον αποδίδει στο κράτος και βεβαίως μπορεί να ε, εκπέσει το ποσό αυτό από τη δήλωσή του και στα δύο καθεστώτα και στις δύο περιπτώσεις ε, εάν ο αποδέκτης ε, είναι καταναλωτής δεν μπορεί να εκπέσει το ΦΠΑ. Γι' αυτό λοιπόν το ΦΠΑ παραμένει ουδέτερο για τους φορολογούμενους και κατόπιν τούτου δεν υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ο αποδέκτης ε, μπορεί να πληρώσει και να εκπέσει το ΦΠΑ και ως εκ τούτου η τροποποίηση αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι ε, μπορεί κατά κάποιον τρόπο να απλουστευτεί η διαδικασία και με τον τρόπο αυτό ε, αποφεύγονται και οι απάτες όταν ο προμηθευτής ε, δεν καταβάλει το ΦΠΑ. Βέβαια, το μειονέκτημα του συστήματος είναι ότι δημιουργούνται άλλοι κίνδυνοι απάτης, διότι το ΦΠΑ τελικά ε, καταβάλλεται στον τελικό κρίκο της αλυσίδας. Κατά την άποψη της Κομισιόν, το σύστημα αυτό πρέπει να περιορίζεται στα γεωργικά και μόνο προϊόντα, τα οποία ε, κανονικά πολλούνται ε, και ε, παρεμβάλλονται μέχρι τον τελικό κατανοητή οι διαμεσολαβητές, οι μεσάντες και πολλοί άλλοι. Πάντως αυτές οι ρυθμίσεις αποκλίνουν από τους ε, κανονικούς ε, κανονισμούς περί ΦΠΑ. Η Ρουμανία πρέπει να λάβει την εξαίρεση από το Συμβούλιο με βάση αυτή την οδηγία και η Κομισιόν εξακολουθεί να εξετάζει το θέμα. Η κυρία Γένσεν. Κύριε Επίτροπε, ε, δεν είμαι σίγουρη ότι σας κατάλαβα. Δεν τα πολύ κατάλαβα. Ε, θα τα εξετάσω εκ των υστέρων. Αλλά ε, το τι μπορεί να γίνει με αυτόν τον νέο κανονισμό για να αποφεύγονται οι απάτες, αυτό που προέκυψε είναι ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα για τους παραγωγούς εκείνους που προέρχονται από άλλη χώρα και έχουν επενδύσει στη Ρουμανία. Εκείνοι δηλαδή οι οποίοι καταβάλουν το ΦΠΑ σε άλλη χώρα και εκεί δεν μπορούν να το εκπέσουν ε, κυρίως όσον αφορά τα έσοδά τους από τη Ρουμανία γιατί δεν έχουν πάρει ΦΠΑ. Η Κομισιόν λοιπόν εξέτασε το πώς μπορεί να επιληθεί αυτό το πρόβλημα για τους παραγωγούς όπως σας είπα από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι όμως έχουν επιχείρηση και στη Ρουμανία και σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να εκπίπτουν το ΦΠΑ με την φορολογική τους δήλωση. Ε, κοιτάξτε, θα ήθελα να πω ότι εξής πρόκειται για ένα νέο μηχανισμό ο οποίος ε, εφαρμόζεται σε διάφορα κρατημέλη παραδείγματος χάρη εφαρμόζεται και στο σύστημα ανταλλαγής ε, ποσοστώσεων εκπομπών. Είναι λοιπόν αλήθεια ότι το σύστημα αυτό προϋποθέτει την καταβολή του ΦΠΑ στο τέλος της αλυσίδας. Αντί δηλαδή να καταβάλει το ΦΠΑ ε, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας. Βεβαίως, βλέποντας τα αιτήματα των κρατών μελών να ε, εφαρμόζεται ένας μηχανισμός αντιστροφής επειδή το ζήτησαν αυτό μέλη, εμείς θα δούμε το θέμα και θα δούμε ε, κατά πόσον υπάρχει στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό λοιπόν και οι προτάσεις ε, της ε, Κομισιόν δεν εφαρμόζονται αυτόματα, ούτε και εμείς τις υποβάλλουμε αυτόματα υποτίθεται ότι έχει προϋπάρξει μια ενδελεχής μελέτη πριν από την ε, κατάθεση της πρότασης. Ε, με τη Ρουμανία συνεργαζόμαστε πάνω από ένα χρόνο ε, για να καταλήξουμε σε κάποια λύση, για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις απάτες ΦΠΑ στα γεωργικά προϊόντα σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι εδώ από την αρχή που αρχίσατε την All και υποτίθεται ότι θα ε, ξεκινάγατε σε 7.30 και υπάρχουν πάρα πολλοί ε, που θα ενδιαφερόντουσαν για την ε, ερώτηση που θα ήθελα να υποβάλω στον κύριο Ρεν. Σας παρακαλώ πολύ, επιτρέψτε μου να κάνω την ερώτησή μου και να απαντήσει η Κομισιόν σε αυτή την ερώτηση. Ο Επίτροπος Υπάρχουν συνάδελφοι που έφυγαν από την αίθουσα γιατί του είπα ότι δεν θα πάρω την ερώτησή του και δεν έχουμε και συμπληρωματική. Είναι δύσκολο και το απόγευμα και συνεχίζεται και δύσκολη βραδιά. Σα είπα μέχρι τι 9 παρατέταρτο θα πάρουμε ερωτήσει. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Πραγματικά ζητώ συγγνώμη, αλλά ε, προσπαθώ ε, να ανταποκριθώ σε όλου του ενδιαφερομένου και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στου επιτρόπου που περιμένουν να απαντήσουν. Τώρα, επόμενη ερώτηση είναι η ερώτηση του κυρίου Παπα-Νικολάου με θέμα τη δήλωση του επικεφαλής του ΟΣΑ για το ενδεχόμενο αναδιάρθρωση του χρέους κρατών μελών της Ευρωζώνης και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ερώτηση απευθύνεται στον Επίτροπο κύριο Ρεν. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, πρόσφατα ε, κλήρωσαν την τρίτη αναθεώρηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας και η κοινή μας γενική εκτίμηση μαζί με την Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό ε, Ταμείο είναι διτή και μπορεί να συνοψιστεί ως εξής. Πρώτον, το πρόγραμμα έχει κάνει περαιτέρω πρόοδος προς τους στόχους του και δεύτερον, απομένουν σημαντικές προκλήσεις να υπερβληθούν για να ε, επέλθει η δημοσιονομική εξυγίανση, να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και ένας βιώσιμος τραπεζικός τομέας. Μπορεί να υπήρξαν καθυστερήσεις σε κάποιους τομείς ή ε, μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για να ε, αποδώσει το πρόγραμμα μέσω πρόθεσμα τίθενται τώρα σε λειτουργία. όλα αυτά θα πρέπει ακόμα να σχεδιαστούν και να επιβληθούν και άλλες μεταρρυθμίσεις για να υπάρξει κριτική, η κρίσιμη μάζα μάλλον για την οικονομική ανάκαμψη και τη βιώσιμη οικονομία. Οι μόνιμες ε, προσπάθειες εξυγίασης του προϋπολογισμού υποστηρίζονται και από ένα τολμηρό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, όπως είπε ο Πρωθυπουργός κύριος Παπανδρέου. Η κυβέρνηση έχει εκφράσει τη δέσμευσή της ε, να επιταχύνει σημαντικά το πρόγραμμα ε, ε, ιδιωτικοποιήσεων για να αποκομίσει 50 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2015 από ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό θα σημαίνει ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα μειωθεί το χρέος ε, κατά 20 και πλέον μονάδες ε, σχέση με το ΕΠ. Επίσης, θα αυξηθεί η οικονομική αποτελεσματικότητα και θα υποστηριχθούν οι μεγαλύτερες επενδύσεις και οι εξαγωγές. Για όλους αυτούς τους λόγους, η πλήρης δέσμευση της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά και η αποφασιστικότητα ε, να αντιμετωπιστούν προνόμια και ε, κατεστημένα συμφέροντα ε, θα είναι κρίσιμα για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι και να αξιοποιηθεί το δυναμικό που υπάρχει για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης των αγορών στην Ελλάδα. Ενθαρρύνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ελλάδα να προχωρήσει στο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησεων. Και αυτό συνδέεται και με την παρατήρηση που έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ. Το 2011 είναι η αποφασιστική χρονιά για την Ελλάδα για να αποκαταστήσει την αξιοπιστία των οικονομικών της πολιτικών και είναι προαπαιτούμενο την Ελλάδα για να ανακτήσει την πρόσβασή της στις αγορές κατά τη διάρκεια του επομένου έτους. Για το σκοπό αυτό οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να επιτύχουν για φέτος το δημοσιονομικό στόχο ή ακόμα και να τον ξεπεράσουν και ε, θα επιτύχουν και τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική τους. Επιπλέον η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει μια αποφασιστική καμπή στις ε, διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις στις επόμενες εβδομάδες και μήνες με αποφασιστικότητα να εφαρμόσει το πρόγραμμα για να ενισχύσει και ε, την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη των πολιτών. Ολοκληρώνω. Είναι μεικτή η στόχη και δημοσιονομική αλλά και το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων πρέπει να εφαρμοστεί. Καθώς επίσης και τα ε, μέτρα ε, αναθεώρησης των τιμών ε, σε σχέση με την αναδιάρθρωση του χρέους θα αντιμετωπιστεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπα-Νικολάου. Κύριε Επίτροπε, πέρυσι συνυπογράψατε ένα μνημόνιο με την Ελλάδα το οποίο προέβλεπε αποπληρωμή του σχετικού δανείου σε 3,5 χρόνια σήμερα εσείς ο ίδιος προτείνετε με δηλώσεις σας επιμήκυνση σε 7 χρόνια που σημαίνει προφανώς ότι κάποιος λάθος υπολογισμός έγινε. Την ίδια στιγμή ο οίκος Moody's υποβαθμίζει αδικαιολόγητα και απαράδεκτα την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε αντίστοιχο επίπεδο με εκείνο της Αγγόλας. Στο τέλος της ημέρας κύριε Επίτροπε Διερωτώμαστε όλοι τι τελικά αρκεί για την ελλάδα για να ορθοποδήσει η απλή επιμήκυνση η μείωση των επιτοκίων που και γι' αυτό έχετε κάνει αναφορές η επαναδιαπραγμάτευση των όρων του μνημονίου το ευρωομόλογο το αναπτυξιακό ευρωπαϊκό ομόλογο όλα τα παραπάνω μαζί μήπως κάτι άλλο μήπως και άλλα μέτρα λιτότητας στην ελλάδα. τι κύριε επίτροπε; Ο Επίτροπος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το βασικό και προαπαιτούμενο και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παραμείνουμε στους στόχους της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με πλήρη αποφασιστικότητα ε, όπως ορίζει το μνημόνιο. Επιπλέον, όπως είπα και στην προηγούμενη απάντησή μου, είναι ουσιώδου σημασίας η Ελλάδα να ξεκινήσει το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο θα βοηθήσει ε, για να μειωθεί το χρέος. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια της συνολικής στρατηγικής που θα αποφασιστεί το Μάρτιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα κοιτάξουν το θέμα αυτό τα κράτη-μέλη της ε, βιωσιμότητας του χρέους και θα ρίνω τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν την επιμήκυνση για τα δάνεια και της Ελλάδας αλλά και να επανεξετάσουν και το θέμα των επιτοκίων των δανείων αυτών. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Και τώρα ερχόμαστε στην ερώτηση που ήταν προς τον κύριο Ντεχόχτ του κυρίου Πόσελτ Αυτό είναι σκέτη φάρσα και αυτό που κάνω τώρα είναι δικαστικό. Μα είπαν στην ώρα των ερωτήσεων ότι θα είναι 7.30 με 8.30. Εσεί ή κάποιο αποφάσισε ε, η καποιο αποφασισε η συζήτηση να καλύψει τον, την ώρα των ερωτήσεων. Είναι από του λίγου τρόπου που έχουμε για να κάνουμε ερωτήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ελλάδα έχουμε κρίση. Οι συνάδελφοί μου, κύριο Μίτσελ και ο κύριο Πάτε Κόπ Κάλαχερ και εγώ έχουμε ερώτηση. Ποιο αποφάσισε. Θέλω να γνωρίζω. Και είναι θεμητή ερώτηση. Ποιος αποφάσισε ότι θα είναι 20 λεπτά οι ερωτήσεις. Και από 20 λεπτά προς κάθε επίτροπο θα γίνουν αυτά 8-9. Ποιος το αποφάσισε. Ακριβώς τώρα θα έκανα μια δήλωση πριν ε, δώσω το λόγο στον Επίτροπο για την τελευταία τελικά ερώτηση της βραδιάς. Και εγώ είμαι εξαγριωμένη και θυμωμένη όπως εσείς, είτε το πιστεύετε είτε όχι. Δεν μου αρέσει να προεδρεύω με τέτοιες συνθήκες και ε, όντω υποχρεωμένη να απογοητεύσω τόσους πολλούς ευρωβουλευτές και να αφήνω τους επιτρόπους να περιμένουν. Πραγματικά θα πρέπει να στραφείτε στους ε, αρχηγούς των ομάδων σας, αν θέλετε ε, να κάνετε τα παράπονά σας, γιατί οι αρχηγοί των ομάδων καθορίζουν την ημερήσια διάταξη και μας εκθέτουν σε τέτοιες συνθήκες σχεδόν σε κάθε εβδομάδα λομέλεια. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να αντιμετωπίσουμε δεόντως και να διεκπαιρεώσουμε τις ε, ερωτήσεις προς το κάθε επίτροπο ή προς το Συμβούλιο. Αυτή η κατάσταση είναι πραγματικά εκνευριστική και απογοητευτική. Το έχω δηλώσει και σε προηγούμενε περιπτώσει. Και όποιο ενδιαφέρεται, παρακαλώ να έρθει σε επαφή με τον αρχηγό του κόμματό του και να εκδηλώσει τα παράπονα και τη διαμαρτυρία του. Γιατί εγώ έχω εγκλωβιστεί στην ημερήσια διάταξη, την... παρακολουθώ την πορεία των εργασιών όπω προβλέπει η ημερήσια διάταξη και δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι, αλλά ποιο αποφάσισε ε, ότι θα γίνουν τρει ερωτήσει προ τον Επίτροπο Σεμέτα και μόνο μία ερώτηση προ τον Επίτροπο Ρεν. Ο κύριο Χίγκιν είχε τη δεύτερη ερώτηση προ τον Επίτροπο Εράν και εγώ την τρίτη. Γιατί ε, ένας Επίτροπος απαντά σε τρει ερωτήσεις και ένα άλλο μόνο σε μία. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Ο κύριο ε, Σεμέτα απάντησε ερώτηση κανονικά του κυρίου ε, ήταν πρώτο στην, ε, σειρά και τώρα θα πρέπει να περάσουμε και στον κύριο Ντεγκούχτ. Πρέπει να, δοθούν απαντήσει από όλου του επιτρόπου. Και ο κύριο Ντεγκούχτ, που είναι ο κύριο Ρεν που είναι πολύ συμβαθή και συνεργάσιμος επίτροπος είμαι βέβαιο ότι βγαίνοντα από την αίθουσα θα έχει την καλοσύνη να απαντήσει και στου τρει σα. Ο κύριο Γκάλαχαρ. Είχαμε τις ερωτήσεις 23 Χιγκής, 24 Μίτσελ και 25 Γκάλαχερ. Εγώ είχα φανταστεί ότι θα απαντούσε ομαδικά στις τρεις ερωτήσεις ο κύριος Ρεν, ο Επίτροπος Ρεν. Γιατί έγινε επιμήκυση της προηγούμενης συζήτησης. Γιατί αυτό γίνεται μονίμως. Όλο βγαίνουμε χαμένοι εμείς στην ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή γιατί παρατείνεται η προηγούμενη συζήτηση. Δεν μπορώ όμως ε, να περάσω και να φάω το χρόνο της επόμενης ε, ολομέρειας που θα αρχίσει σε νέα. Είχα υποσχεθεί στον κύριο Πόσολ και στην κυρία Τσικάου να απαντηθούν οι δικές τους ερωτήσεις. Και κανονικά οι τρει δικέ σα θα ήταν οι τελευταίε αν είχαμε προχωρήσει με ταχύτερου ρυθμού, αλλά δυστυχώ δεν προλάβαμε. Αυτή τη φορά τελικά έτσι πω καθυστερήσαμε δεν μπορώ καν να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Πόσελτ. Λυπούμε ειλικρινά, δεν λυπούμε απλώ, αλλά είμαι και εξοργισμένη. Αλλά είδατε τι συνέβη όλη τη μέρα με την ημερήσια διάταξη. Και πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστη αυτή η κατάσταση. Επιτρέψτε μου λοιπόν, όπω είπα, να περάσουμε προ την ερώτηση προ τον Επίτροπο Ντεγούχτ που θα απαντήσει ο κύριος Σεμέτα που τον αντικαθιστά και όπως είπα θα είναι η τελευταία ερώτηση της βραδιάς δυστυχώς. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε, και λυπούμε που γίνατε σε αυτών των εσωτερικών δυσκολιών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση είχε ε, αρνητικό αντίκτυπο στο διμερέ εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Ανατολικής εταιρική σχέση. Μόνο με, μεταξύ του 2008 και του 2010 είχαμε μείωση του εμπορίου αυτού κατά 20%. Η ανατολική εταιρική σχέση άρχισε να εφαρμόζεται όσο μεσουρανούσε δυστυχώς η χρηματοπιστωτική κρίση. Και μάλιστα είχαμε τη διάσκεψη κορυφή 7 Μαΐου του 2009 Είχαμε βέβαια κάποιες ε, ε, δημιουργίες ε, δομών και κάποιες πολυμερείς πλατφόρμες. Η εταιρική όμως ανατολική σχέση ήταν στα σπαργανά της και δεν μπόρεσε να ελαφρύνει ή να αποδυναμώσει τις αρνητικές συνέπειες παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Δυστυχώς δεν υπήρχε συνέργεια σε θέματα ανατολικής εταιρικής σχέσης και ε, η στρατηγική για τον εύξηνο πόντο είναι θέμα πολιτικό περισσότερο και όχι τόσο εμπορικό οικονομικό. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στον Νότιο Κάφκασο δεν είχε, δεν είχε επιρροή στη, στο εξωτερικό εμπόριο και οι προετοιμασίες για νέα συνεργασία, και μια νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου διεξάγονται με την Αρμενία και τη Γεωργία. Ενώ η είχαμε συμφωνία εμπορική σχέση με το Αζερβαϊτζάν που αυτή τη στιγμή τη χάνουν κάποιε αναβάθμισει. Σα ευχαριστώ, κύριο Πόσελτ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την τόσο ακριβή απάντηση. Πολύ σύντομα, διαβλέπετε καμία δυνατότητα για ε, εντατικοποίηση του εμπορίου με τις χώρες του Νοτιού Καυκάσου βοηθώντας να αποκλιμακωθεί η ένταση εκεί και ιδιαίτερα και σε σχέση με την εξωτερική πολιτική σε θέματα ενέργειας της Ένωσης. Ο Ευχαριστώ. Όπως είπα και στην απάντησή μου, μας απασχολεί το θέμα ε, μιας ε, γενικευμένης ζώνης ελεύθερου εμπορίου και βαθιάς, ε, εμβριθέστερης και θα υποβάλουμε τις, ε, τους βασικούς προσανατολισμούς και τις συστάσεις προς τις χώρες για να δούμε τι χρειάζεται για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τέτοιου είδους ευρυθέστερες ε, και ευρύτερες εμπορικές σχέσεις. Οι συμφωνίες αυτές θα προχωρήσουν αν οι ενδιαφερόμενες χώρες ε, κάνουν εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους. Γιατί μερικές το θέλουν και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντικοποίηση του εμπορίου με τις χώρες αυτές. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρλι. Πρόλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Περίμενα να τελειώσετε το χρόνο των ερωτήσεων πριν σας διακόψω, γιατί ξέρω ότι δεν είχαμε χρόνο. Αλλά εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοί μου, θα θέλαμε να γραφεί στα πρακτικά της Ολομέλειας ότι αυτό είναι μια επιπλέον αποδυνάμωση ε, βασικού ε, εργαλείου που έχουν οι βουλευτές εδώ και μάλιστα των ορεινών εδράνων. Καταλαβαίνω ότι θέση σας, αλλά αντίστοιχα δεν φταίνε μόνο οι αρχηγοί των πολιτικών ομάδων, γιατί ε, η διεξαγωγή των εργασιών είναι θέμα Προέδρου. Και αυτός που προείδρευσε πριν από εσά άφησε τα πράγματα να εξοκύλουν τόσο πολύ. Δεν ξέρω, ίσως θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε εσεί στο Προεδρείο, να το δείτε μεταξύ σα, οι Αντιπρόεδροι και να συμφωνήσετε ότι αυτό το τμήμα, ω ώρα των ερωτήσεων είναι ε, ιερό και απαραβίαστο και όταν ε, δεν μπορούν κάποιοι να ολοκληρώσουν τα θέματά τους να το διακόπτουν για την ώρα των ερωτήσεων. Θα το θέσω υπόψη και εγώ του Προέδρου της ομάδας μου αλλά και εσείς παρακαλώ στο Προεδρείο. Ευχαριστώ κύριε Κρόλη. Θα το θέσω υπόψη των Προέδρων των πολιτικών ομάδων γιατί λυπούμε πολύ αλλά αυτό είναι εκεί η διάσκεψη των Προέδρων όταν ορίζει την ημερήσια διάταξη. Φορτώνει πάρα πολύ την ημερήσια διάταξη πριν φτάσουμε στην ώρα των ερωτήσεων. Και έχετε δίκιο ότι κάπως πρέπει να ε, τερματιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτή η ώρα των ερωτήσεων πραγματικά που ε, λογοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους βουλευτές και το Συμβούλιο θα πρέπει να ε, είναι εξασφαλισμένη. Και αύριο το πρωί το πρώτο πράγμα που θα γράψει στον υπολογιστή μου θα είναι αυτό, να είστε βέβαιος. κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πριν από λίγο είχατε υποσχεθεί ότι θα δινόταν απάντηση και στη δική μου ερώτηση από τον, κύριο, από τον Επίτροπο έχω αλλά βλέπω ότι έφυγε ο αρμόδιος Επίτροπος. Εγώ όμως περιμένω την απάντησή μου. Νομίζω ότι σήμερα καταπατήθηκαν όλες οι διαδικασίες. Δεν έγινε σεβαστό τίποτα και πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς ξέφυγε έτσι η κατάσταση. Κυρία Τσικάου, εγώ είχα την καλή πρόθεση να απαντηθεί και η δική σας ερώτηση. Αλλά εξαιτία πίεση χρόνου και επειδή έπρεπε οπωσδήποτε να σταματήσουμε σε 9 παρατέταρτο, δυστυχώ φτάσαμε σε 9 παρατέταρτο πριν προλάβουμε να ακούσουμε και την απάντηση στη δική σας ερώτηση. Ούτε και εμένα μου αρέσει αυτή η κατάσταση. Είμαι πολύ δυσαρεστημένη με αυτά που έγιναν, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο για να διεκπαιρεώσουμε περισσότερες ερωτήσεις. Έκανα ό,τι μπορούσα. Είπα συμπληρωματικέ μόνο από τους τάκτες των ερωτήσεων, σε κανέναν άλλον. Αλλά παρόλα αυτά δεν καταφέραμε εγκαίρως να φτάσουμε και στη δική σας ερώτηση. Δεν ήταν μόνο η δική ερώτηση που δεν απαντήθηκε, αλλά όλες όσες ερωτήσεις έμειναν απάντητες θα απαντηθούν γραπτώς. Ολοκληρώνεται η ώρα των ερωτήσεων τώρα και ευχαριστώ τους διερμηνείς και το προσωπικό για την ανοχή τους. Η συνέχεια της Ολομέρης 9.